So, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ για να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Und es geht jetzt weiter in den Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το σημείο 10, τροποποίηση της οδηγίας για την ποιότητα των καυσίμων και την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, έμεση αλλαγή χρήσης γης και κατόπιν θα ψηφίσουμε το σημείο 11, τροποποίηση της οδηγίας για την αξιολόγηση των ε, δημοσίων και ιδιωτικών έργων για το περιβάλλον, αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επειδή είναι αρκετή ψηφοφορία, σας παρακαλώ να είστε λίγο πειθαρχημένοι, δεν έχουν έρθει όλοι οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να κάνουμε έναν έλεγχο, να δείτε αν έχετε τις ηλεκτρονικές σας κάρτες, διότι χωρίς κάρτα δεν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε την ψηφοφορία. Δεν μπορώ να κάνω καμία εξαίρεση. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την έκθεση της κυρίας Λεπάζου. Είστε έτοιμοι. Να ξεκινήσουμε. 226 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 317 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τώρα, 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση δεν ήταν σαφές. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 29 προς 19 εγκρίνεται. 19 υπέρ. κατά απόχες εγκρίνεται 227 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται 228 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται τραν 18 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται η Consolidated 4 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Ενοποιημένη 1 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική 3 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 245 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Dann geht's weiter mit 208 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές Είναι Ενοποιημένη από τα υπέρ. Κατά αποχές. Α το ελέγξουμε καλύτερα αυτό ηλεκτρονικά. Ενοποιημένη από τα... Haben alle. Alde hat einen zu viel in der Abstimmung. Jetzt ist in Ordnung. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. 200 und Εγκρίθηκε. 257 είπε. κατα Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 259-60 και άκρη 20 ταυτίζονται και ψηφίζονται και μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τσεκ! Ηλεκτρονικά λοιπόν και τις τρεις αυτές αρχίζει. Ψηφίσατε. Πέρας. Απορρίπτονται. Ήτρε 23 ψηφίπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. ITRE 23. Ηλεκτρονικό έλεγχο θέλετε για την 23 της Επιτροπής Βιομηχανίας μάλιστα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 24 η τρύπε. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 62 π Κατά. Αποχές. Απόρριψτε. Η Η35Π. π Κατά. Άποχες έλεγχος. Για την 25 της ήτρε, παρακαλώ, ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. Είναι τα 13 υπέρ. Dagegen. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας το λέξουμε για καλό και για κακό. Είναι τα 14 ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ist Εγκρίνεται. Είναι τα 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Είναι τα 16 υπέρ. Dagegen. Κατά. Enthaltung. Wir Αποχές. Ας το ελέγξουμε. Είναι τα 16 παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είναι κρίθηκε. 264 επέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 265 επέ. Κατά. Αποχές επίσης εγκρίνεται. 266. Επιθυμεί κάποιος τσεκ. Ωραία, ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά τη 265 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 266 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 268 και δεύτερο 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και εδώ κάνουμε ένα άλμα και πάμε στην 27. Μικρόμεν υπέρ ε, κατά αποχές Νομίζω ότι έχει εγκριθεί, αλλά καλύτερα στο ελέγξουμε παρακαλώ για την 27. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είναι σαφέστατα εγκρίθηκε. 273 υπέρ. Κατά αποχές που ε, απορρίπτεται. Τραν 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 274, 275 και άγρι 22. Ομού υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τι θέλουμε, έλεγχο για την 30, παρακαλώ, ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Σαφές δεν είναι. Γιατί θέλετε έλεγχο. 284, 285, 286. Υπέρ. Dagegen. Κατά. Αποχές. Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το σύνολο. Εντάξει. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist Α, Απορρίπτεται. 287 ε, και αγρί 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 288 και τράν 23 μαζί υπέρ κατά Το ΕΛΚ γιατί δεν ψηφίζει, μπορείτε να με εξηγήσετε. Έλεγχος παρακαλώ. Είναι πολύ... So, haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. Δύο ενενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. 2.93 υπέρ κατά Απορρίπτει 2,94 και άκρη 25 Είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, δύο, συγγνώμη, 96, διορθώνει ο πρόεδρος γιατί είχε πει 2,66. 2,96 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η άγρη 26 καταπίπτει και συνεχίζουμε με την 300 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 304 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε μέσω τώρα στην ενοποιημένη 6 υπέρ. κατά άποχες ας λέξουμε καλύτερα ενοποιημένη έξι παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται η 308 είπε κατά αποχές απορρίπτεται 310 3π κατά αποχές απορρίπτεται 309 και η 329 επέ κατά αποχές απορρίπτεται η 33 επέ κατά αποχές εγκρίνεται 34 επέ κατά εποχές εγκρίνεται 35 επέ κατά εποχές εγκρίνεται 36 επέ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 312 και άκρη 30 υπέρ κατά αποχές απορρίψεται. 313 και τράν 27 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφέ, στο το ελέγξουμε παρακαλώ. Haben alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Ψηφίσατε όλοι, βέβαια. Απορρίπτεται. Τρία και άκρη τριάντα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία δεκαεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 318 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε παρακάτω άγκρι 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται είναι τα 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τραν 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεβέ 20 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα. Να το λέξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Δεβέ 20. Ψηφίσατε όλοι. Επέρας. Ε, γι' αυτό δεν κατάλαβα. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος. Έχουμε την ενοποιημένη 5 προηγουμένως. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.40 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τη 40 της Επιτροπής Γεωργίας υπέρ, άγκρι 40, κατά, αποχές απορρίπτεται, άγκρι 41 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 404 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι σαφές. Ε, ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 46 παρακαλώ. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ist angenommen. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τη 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Α, θέλετε έλεγχο. Καλώς. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 47 παρακαλώ. Haben alle abgestimmt? S und D. Ψηφίσατε όλοι. Σοσιαλιστές και δημοκράτες, ένας υπεράριθμος. Τώρα είναι εντάξει. Εγκρίνεται. Ή 334 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 405 και άκρη 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφτεται. 406 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται είναι τα 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 409 είναι τα 23 θέλετε έλεγχο όχι κατά λάθος σου ζητήσατε όχι, τσεκ. Μάλιστα. Okay, es Ας την ελέξουμε. Είναι τα 23 λοιπόν. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασα. κρίνεται λοιπόν. Η 409 επέ. Κατά. Όποχες απορρίπτεται. 49 επέ. κατά αποχές εγκρίνεται. 410 και ντεβε 24 δεν χρειάζεται να ψηφιστούν. Άλμα τώρα στο κείμενο. Ψηφίζουμε 418, 19 και άγκρι 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται. Τσεκ φωνάζει κάποιος από κάτω. Ωραία. Ας το ελέγξουμε τότε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψτε. 424 υπέρ κατά αποχές. Ich wiederhole es nochmal. Επαναλαμβάνω. 424. Ψηφί υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, τώρα αυτό θέλει έλεγχο, λέει η κυρία Κλάσσο. Ψηφίσατε όλοι. 4.24. Και στα αγγλικά. Ψηφίσατε όλοι. Βέβαια. Εγκρίνεται. Είτε 35 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τσακ. Για την Ήτρη 35, ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλα. Πέρασε. Απορρίπτεται. Ήτρη 36, είπε. Κατά. Αποχές. 4.21 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ενοποιημένη 10 είπε κατά αποχές εγκρίνεται. 422 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. 425 τραν και άγκρι είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. Άκρη 47 είπε, Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4, 27 είναι τα 27 μαζί. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 428 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Είναι τα 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απόρριψετε. Είναι τα 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 4.30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4.31 υπέρ. Dagegen κατά αποχές απορρίπτεται 432 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ήρθε 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 434 και 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται για κάνε ένα έλεγχο, λέει η κυρία Κλάς. Μάλιστα. 4.34 και 28 κατόπιν αιτήματό σα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Αγκρίθηκε. Ah, jetzt geht's weiter mit 56 dafür. <laughs> Υπέρ της επόμενης 56 κατά αποχές εγκρίνεται. 4.39 και άγκρι 49 μαζί. είπε. Κατά αποχές απόρριψετε. 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 58. Τι θέλετε έλεγχο για την 57 ωραία. Ηλεκτρονική απολύθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Εγκρίθηκε. 58 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59 είπε. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 59 για καλό και για κακό. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 4.46 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 60. Τι θέλει έλεγχο 60. Όχι καταπίπτει. 4.47, ε, 4.48 και άγκρι 51. Ψηφιπέ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 449 τραν 38 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε 451 και άγκρι 52 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίψετε Θέλουμε έλεγχο γι' αυτό. 4.51 και άγκρι 52. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απερίφθησαν. Τώρα, τραν 40, υπέρ. Τραν 40, υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίψτε. Η 457 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 341 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άλμα τώρα. 480. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφής. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά 480. Ψηφίσατε όλοι πέρας. συγκρίθηκε. 481 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 57 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 482 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα το παράρτημα. Πρώτον, 484 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 488 και 489 και άκρη 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 490 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 492 υπέρ κατά αποχές απορρίψετε. Η 65, 493 μαζί υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε παλήθευση αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίω. Αρχίζει τώρα για την 65 και την 493 ψηφίσατε όλοι πέρα. Εγκρίθηκαν. 66 και 4,91 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές, σας θα ελέγξουμε παρακαλώ και αυτό ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. 37 υπέρ, 32 κατά, εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τσεκ για την 4-6 παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση. Αφού το ζητάτε ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απόρριψετε. und DB30 dafür. DB30 και 67 υπέρ Κατά αποχές 499 είπε. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. Κάποιο ζήτησε τσεκ για, για την 499. Λοιπόν, ας το ελέγξουμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρασε. Es Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε, αλλά δεν σηκώνεται χέρια. Εγώ πού να το καταλάβω ότι είχε εγκριθεί. Μήπως να μας φέρουν τον καφέ για να πάρουμε λίγο μπρος. 503, 504, 505, Ήτρε 43 ε, και Άγκρη 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 506 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 507 και Ρέγγι 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 508 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 509 επέ, κατά αποχές εγκρίνεται. das mal elektronisch. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Abgestimmt. Ψηφίσατε όλοι. Βέβαια. Ist abgelehnt. Απορρίπτεται. 70 και 510. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ή μήπως όχι. Καλύτερα να το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κάποιος δεν μπορεί να μας φέρει λίγο καφέ για να είμαστε και στη θέση να ψηφίσουμε. Θα ε, ανοίχατε την καλοσύνη. 5-15 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος γιατί 5-15. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. 517 καταπίπτει. Και συνεχίζουμε με την 72, DV32 και ΙΝΤΑ 33. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 518 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Wir machen Συνεχίζουμε. Είναι τα ένα. Τα βρήκατε στους καταλόγους ψηφοφορίας σας. Είναι τα ένα. Είναι σε αιτιολογικές αναφορές και σε μένα στη σελίδα 40. Citations. Αιτιολογικές αναφορές. είπε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τραν 1. είπε, Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η αγκρίανα υπέρ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84. 80 geht's weiter. όχι, 86. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ε, να έχουμε παρακαλώ την 86 ηλεκτρονικά. Ψηφίζετε όλοι. ένας. Εγκρίνεται. 87 και άγκρι 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Είναι 92 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94. Τι θέλετε, έλεγχο για την 92 και την Ήτρε 2, παρακαλώ. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen und somit ab. απορρίπτεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η άκρη 4 καταπίπτει, 93 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Αποχέ. Συγγνώμη, κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρεγγένα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 99 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλα. Πέρασε. Αμάν. Αμάν τι σηκώνετε χέρια, τι να κάνω κι εγώ. Ε, η τριτρία. Υπέρ, ε, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100, 101, 102, 103, 104 και άγκρι 7. Ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές, δεν είναι σαφές, για καλό και για κακό, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η επαλήθευση. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist Ψηφίσατε Ist abgelehnt, der Block. 108. Απορρίπτεται. 108 ψήφι υπέρ. Α, περιμένω. 108 dafür. Dagegen. 108 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύε 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 116 πε. κατα Κατά. Απορρίπτεται. ΔΒ5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με τη Τζούλι Γκέρλινγκ, 136. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 138. Την ψηφίζουμε. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ελέγχουμε την ίντα 3. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρεκί 5 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφέ Ας το ελέγξουμε παρακαλώ. Είναι η πέντε της περιφερειακής ρέγγιφου. Ε, 5. Ψήφισατε όλοι. Πέρα. Απορρίπτεται. Είναι τα τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρεγγί 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 5 και τράνε 7 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Είναι τα 5 και τράνε 7 μαζί. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ist klar abgelehnt. Απορρίπτεται σαφέστατα. Συνεχίζουμε. 177. Υπέρ. Κατά. Είναι της κυρίας Βίλης τροπολογία. Αποχές. Δεν ψηφίζετε παρακαλώ, ας το ελέγξουμε. 177 ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Γκρίνεται. ΔΕΒΕ 10 καταπίπτει και προχωρούμε. Μια στιγμή να δω που θα πάμε τώρα. ΔΕΒΕ 11 είπε. Κατά αποχές εγκρίνεται. Εκατόν Βίλς είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ας την ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά καλύτερα. 186 της κυρίας Βίλς. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Όχι, εγκρίνεται. Δώδεκα υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφής. Ας το ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 13. Απέ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αλλά ας το επαληθεύσουμε. Δεν σηκώνετε χέρια δυστυχώς. 13. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Ζιλ Παρνιό. 185, Ήτρε 15 και Τραν 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 202. Υπέρ. αυτά. αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 202 παρακαλώ ψηφίσατε όλοι πέρας απορρίψατε η 203 Παναγιώτοφ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 14 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση για την 14 της ΔΕΒΕ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ingredient 206 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 207. 208 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. η 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με τη Ρέγγι 11 στην τελευταία σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 321 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.25 υπέρ Κατά. Αποχές απορρίψετε. Ραγή 12 ειπέ. Κατά. Αποχές απορρίψετε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. 43 υπέρ, 26 κατά, μία αποχή. Και η δεύτερη ηλεκτρονική υποφορία για το νομοθετικό ψήφισμα αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 43 υπέρ, 26 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία εισηγήτρια. Σας δίνω και το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να ευχαριστήσω διότι επέδειξαν πνεύμα συνεργασίας ε, στη διάρκεια όλων των εργασιών ε, κατά την προετοιμασία των ε, τροπολογιών παρά το γεγονός ότι στο τέλος δυστυχώς ε, δεν υπερψήφισαν όλη αυτή την έκθεση και θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως ε, τη ε, ομάδες της Επιτροπής ΕΜΒΗ, των Φιλελευθέρων και τους δικούς μου τους συνεργάτες, διότι εργάστηκαν και πολλές ώρες σε αυτό το δύσκολο κείμενο. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό για να προετοιμαστούμε για την Ολομέλεια. Ευχαριστώ όλους. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια από πλευρά μου ξανά και προς τους συνεργάτες, το προσωπικό και τη γραμματεία. Ήταν μακροσκελέστατος ο κατάλογος ψηφοφορίας και χρειάστηκαν και συμβιβασμοί. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht des Kollegen Andrea Τώρα έχουμε την έκθεση του συνάδελφου Αντρέα Τζανόνι. Και είστε όλοι εγκάρδια προσκεκλημένοι να συνεχίσετε να ψηφίζετε. Και όλοι οι υπόλοιποι παρακαλούνται να ηρεμήσουν γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ψηφίζουμε σε τέτοιες συνθήκες θορύβου. Αρχίζουμε. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 111 υπέρ και η 12 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Θέλετε έλεγχο για την 111 και 112 παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 34 υπέρ, 32 κατά. Εγκρίνεται, συνεπώς. 113 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 114. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 116 π. Κατά. Έλεγχος. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. 116. Ψηφίσατε όλοι. Φέρες. Απορρίψατε. 117 επέ Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 είπε. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε τα 119 ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ας το αλλάξουμε καλύτερα. 120. 120. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Κανονικά με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Τι αρμονία είναι αυτή. Ε, ενοποιημένη έξι. Υπέρ. Κατά. Μόνο οι πράσινοι ψηφίζουν. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ ψηφίστε. Δεν μπορώ να σας βλέπω. Αμαντεύω μαντεύω τι θα ψηφίσετε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 121 είπε. Κατά. Λοιπόν, και πάρει ηλεκτρονικά. Όσο δεν σηκώνετε χέρια θα ψηφίζουμε μία-μία ηλεκτρονικά άμα θέλετε. Μπορώ και έτσι. Ε, ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124, 125 και 5, 23 υπέρ κατά δεν είναι σαφές ηλεκτρονική επαλήθευση. Haben alle Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 522 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η τραν 5 υπέρ, Κατά. Έλεγχος. Τραν πέντε. Ψηφίσατε τώρα, Πέρας. Εγκρίνεται. 521. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 Κατά τμήματα, παρακαλώ. Τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές, ναι. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 158. Υπέρ. κατά αποχές Συγκρίνεται. 189. Ναι, επέ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Δεν τα βλέπω. Ε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 189. Ψηφίσατε όλοι. Βεβαίως. Εγκρίθηκε. Η ενωπημένη 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, ελέγχουμε την ενωπημένη 7. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 199 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Η συμβιβαστική 8. Πώς είπατε? Θέλετε έλεγχο 199 ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλιστα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Jetzt geht's weiter mit Abänderungsantrag 200. Συνεχίζουμε 222. Το δεύτερο τμήμα όμω. Δεν σα λέω πια οι σελίδες από χτες. 222 δεύτερο τμήμα άρθρο 1 σημείο 4. Σε μένα σελίδα 11. 222. Εσείς έχετε άλλες σελίδες, μου το είπατε χτες. 222. Ε, Α, 220 διορθώνει ο πρόεδρος τώρα. 220. Το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Τώρα συμφωνήσαμε, τα βρήκαμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Συμβαστική 8, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Consolidated 9. Dafür. Η ενοποιημένη 9. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τραν 13. Τραν 13. Στο δικό μου κείμενο σελίδα 20. Τραν 13 είπε. Κατά. Αποχές. Άλλα ντάλλον. Λοιπόν, ας ε, ε, ε παρθέψουμε ηλεκτρονικά τη 13. Πέρας ε, εγκρίθηκε σαφώς. 3.33 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε 3.34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Σας ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά την 3.34 αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Βέβαια. Εγκρίνεται. 3.35 πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 πέρα. Κατά αποχές. Περιπτέται. 3.36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.37 339π Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.39 πέρ. Αυτά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ την 3.39. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται η ισοψηφία. 3.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 3.41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 344 και 45 μαζί. Είπε, Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 346 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 347 υπέρ. Α, και 543 μαζί. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για αυτές τις δύο. 347 και 43 των αναφορών. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Εγκρίθηκαν με σαφή διαφορά. 348 υπέρ. Κατά. Εποχές. Έλεγχος. Εδώ δεν συμφωνούμε. 348, ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. 542 και 44 υπέρ. Τελείωσε η προηγούμενη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 349 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Ορίστε, θα ελέγξουμε την 349 ζητάτε μάλιστα. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίνεται. Η 350 καταπίπτει, ενωπημένη 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 411 της κυρίας Τάισεν. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4-12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 413 υπέρ κατά αποχές ας το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά είμαστε στην 413 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 4, 21, 4, 22, 4, 23. Επόμενη σελίδα στη δική μου λίστα υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτωται. 39 υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5.50 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ασαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 50 της Επιτροπής Αφόρων. Ψηφίσατε όλο. Πέρα. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ωραία. Ηλεκτρονικά. Την 424. Ψήφισετε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 425. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 427 και 552 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 408 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 429 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 430 επε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 431 επε Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 432 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 433 επέ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 44 και 35 Είπε. κατά αποχές απορρίπτεται. 4, 36, 37, 38, 39 και 40 και 5, 53 όλες αυτές μαζί Είπε. κατά αποχές απορρίπτονται. 20 το μεταφορών είπε. αποχές απορρίπτεται. Τραν 21 υπέρ 100. αποχές απορρίπτεται. 441 υπέρ 100. αποχές εγκρίνεται. 442 υπέρ Θέλετε παλήθευση. 442. <laughs> 442 dafür. επέ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 47 επέ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 443 υπέρ. Dagegen. Haltung ist... Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 444 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. 445 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 454 υπέρ κατά αποχές δεν κατάλαβα ψηφίζουμε την 454 ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα η σοφορία. ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίθηκε Πάμε στα παραρτήματα πλέον. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αλλά στο έλεξουμε καλύτερα. 49. Παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση γιατί δεν ήταν σαφές. 49. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε. 5.54 54 είπε. Δεν σηκώνεται χέρια. 5.54 54 ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Ναι, προφανώς τώρα ναι. Γκρίνεται σαφώς. 456 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 457 υπέρ. Κατά. Αποχές. 457 ηλεκτρονική überprüfung. 457 ηλεκτρονική επαλήθευση. Haben alle abgestimmt und auch richtig. Ψηφίσατε όλοι και σωστά ελπίζω όλοι. Πέρας. Δεν Ευχαριστώ πολύ. 50. το εισηγητή. Σε πολλά τμήματα. Τρία. Θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Τμήμα πρώτον. Αρχίζει η ψηφοφορία υπέρ. Να το κάνουμε καλύτερα ηλεκτρονικά από την αρχή. Ωραία. Το πρώτο τμήμα ηλεκτρονικό. 50. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται το πρώτο τμήμα. Έτσι. Τμήμα δεύτερον. Και πάλι ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Και αυτό εγκρίνεται. Και πάμε στο τρίτο τμήμα. Και πάλι ηλεκτρονικά αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίθηκε και αυτό το τμήμα. Es Πάμε αμέσως τώρα στην 465. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 466 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 467 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται. 468 είπε. κατά αποχές εγκρίνεται. 469 είπε. τσεκ άμα θέλετε θέλετε 468 τότε. Έχει ζητήθει ηλεκτρονική επαλήθευση, ψηφίσατε όλοι. Φέρας. Εγκρίθηκε. 469 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 69, έλεγχος. Ελέγξτε το. Έλεγχος. 469. Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκε. 11 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Γενοποιημένη 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Als nächstes stimmen wir über 543. Πάμε στην 543. Ψηφί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5.44 υπέρ ε, κατά αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, φωνάζει κάποιος από κάτω. Για την 5.44 στην ελέξουμε. Λοιπόν, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Εγκρίνεται. Με υψηλό ψηφία αρκετή. Η ενοποιημένη 13, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε σε τελογικές σκέψεις τώρα, recitals. Πέτη 1. ψηφί πέ, στην πρώτη τελογική σκέψη. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62, Επέ. Κατά, Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 62 παρακαλω Ψήφισα τέλη. όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 5-2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ. συγκρίθηκε. Καλώς. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 67. Αρχίζει τώρα ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα. Ist klar angenommen. Damit fällt Petit 4 und wir machen weiter mit Petit 5. Καταπίπτει 4, 5, 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 και 69. Ταυτίζονται υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 7 υπέρ. Dagegen. Haltung ist Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, δεν είμαι σίγουρος. Δεν είδα καλά. Ας ελέγξουμε παρακαλώ την πέτη 7 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Το ε, Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 5 8 είπε. Dagegen, Haltung ist angenommen. Κατά αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 5 9 κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 77 είπε. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 78 είπε. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση και πάλι. Παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίθηκε. 79 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ενοποιημένη 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ το 85. Ψηφίσατε. όλοι. Πέρα. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Ενοποιημένοι 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 90 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ψηφίζουμε την 88 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Πέρασε είπα, <laughs> δεν κλείνει. Α, απορρίπτεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. Η 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ελέγχουμε την 513. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίψετε. 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 514 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 515 δεν ψηφίζεται μου λέγουν. Τραν λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Υπτά. Τσεκ. Μάλιστα γιατί είναι 91 ηλεκτρονική επαλήθευση αφού το ζητάτε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Η 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Για να το ελέγξουμε παρακαλώ ηλεκτρονικά αυτό. Τραν 3. Ψήφισατε όλοι. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. Οκτώ κατά τμήματα, δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Κάντε υπομονή σας παρακαλώ, μισό λεπτό, κάνουμε έλεγχο, μην κάνουμε κανένα λάθο και χρειαστούμε καλοκαιριάτικα να ξαναγυρίσουμε να ψηφίζουμε εδώ πέρα. Hm? No problem. Συνεχίζουμε στην τελευταία σελίδα, τραν 4 στη δική μου λίστα, υπέρ. Κατά. Αποχές, δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Stimmt. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, δέκα, έντεκα, υπέρ κατά αποχές υπέρ τη 17 υπέρ εγκρίθηκαν οι προηγούμενοι ε, κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την υπέρ τη 17 ψήφισατε όλοι πέρας απορρίπτεται λοιπόν φτάσαμε στην τελική ψηφοφορία εσείως η πρώτη είναι τώρα το σχέδιο της έκθεσης Ψηφίζετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνετε; Το δεύτερη ηλεκτρονική ψηφοφορία, το νομοθετικό ψήφισμα, ανοίγει τώρα, αρχίζει. Ψηφίζετε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται επίσης με μεγάλη πλειοψηφία. Και απευθύνομαι στον εισηγητή. Κύριε Τζανόνη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους, ευχαριστώ τους και εισηγητές, ευχαριστώ τη Γραμματεία της Επιτροπής Περιβάλλοντος, τη Γραμματεία των Φιλελευθέρων και όλο το προσωπικό που συνεργάστηκε μαζί μου. Ήταν πολύ καλή δουλειά, καταλήξαμε σε συμβιβασμούς ε, και σε κάποιες συμφωνίες, αλλά... Νομίζω ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να εφαρμόσουμε τη διαδικασία του άρθρου 70, επομένως θα πρέπει να πάμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Äh, είναι σαφές λοιπόν. Δεν θα ψηφίσουμε για τη χορήγηση εντολής ε, διαπραγματευτικής. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σας συγχαρώ. Σωστά δεν τα λέω. Ε, συγχαρητήρια. Θα πάμε στην Ολομέλεια. Δεν θα ψηφίσουμε εδώ για τη διαπραγματευτική εντολή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη γραμματεία και τον ε, γραμματεία τον κύριο Εμιλιάνο. Θα τα ξαναπούμε το απόγευμα, μην μου φύγετε. Έχουμε Υπουργό Υγείας. Για τους ε, ελαχίστους που θα αποσιάσουν το απόγευμα, να ευχηθώ καλές διακοπές, να φορτώσετε τις μπαταρίες σας με ενέργεια και να ξανάρθετε μετά το καλοκαίρι. 11 η ώρα και 30 συνεδριάζουν οι συντονιστές, 11.30 συντονιστές.